η προσωρινή η προφορική ερώτηση για τις διαπραγματεύσεις υπό την του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού όσον αφορά την ασφαλή και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων. Έχουμε μείνει 10 λεπτά πίσω στο χρόνο, οπότε πρώτα απ' όλα τον λόγο έχει ο κύριος Μπλόκλαντ για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, Ολομέλεια πέρυσι τον Μάιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια πολύ σαφή θέση όσον αφορά το αρνητικές επιπτώσεις της διάλυσης πλοίων στην ε, Ασία, τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει αυτή στο περιβάλλον καθώς αυτά τα πλοία διαλύονται επί της ακτής και η ανακύκλωση αυτή η οποία γίνεται δεν είναι τόσο φιλική προς το περιβάλλον. Στον Παγκλαντές παραδείγματος χάρη υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία όπου γίνεται διάλυση των πλοίων και δεν είναι η πιο φιλική στο περιβάλλον. Όμως το ΔΕΚ ε, εξέδωσε μία απόφαση σχετικά και τα δικαστήρια του Μαγκλαντές, με συγχωρείτε, πως έπρεπε να κλείσουν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις των Μπαγκλαντές και οι αρχές εκεί θα πρέπει εντός τριών μηνών να βρουν μια λύση η οποία θα πληρεί τις ε, προδιαγραφές συμφωνίας της Βασιλείας. Αυτά αναφέρονταν και στο κείμενο το οποίο ενέκρινε πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως, δεν ξέρω, το δικαστήριο στο Μαγκλαντές διάβασε την έκθεσή μας. Οπωσδήποτε είναι μια απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση για αυτές τις ε, πρακτικές. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ένα δικαστήριο στο Μπαγκλαντές και σε άλλες χώρες της ε, Ασίας ε, έλαβε τέτοια απόφαση. Προφανώς οι χώρες δεν ε, κάνουν αρκετά και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Το Μάιο στο Χονγκ Κόνγκ θα, θα γίνει μια παγκόσμια διάσκεψη υπό την αιγύδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με αντικείμενο να επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία για την ανακύκλωση των πλοίων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος οφείλει να διασφαλίσει πως το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα στείλει ένα σαφές μήνυμα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτή τη διάσκεψη υπό το φως των όσων ακούστηκαν πέρσι και θεωρώ πως θα πρέπει να προσθέσω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, επικίνδυνες ουσίες ε, οι οποίες μεταφέρονται από ένα πλοίο ή υπάρχουν σε ένα πλοίο μπορούν να θεωρηθούν πράγματι ουσίες που καλύπτονται από την συνθήκη της Βασιλείας. Η τροπολογία υπερθμών 1 του ΕΛΚ εξασθενεί την σχετική ε, διάταξη. Εάν τα πλοία διαλύονται στην ε, ακτή, ε, αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Πρέπει λοιπόν πριν περάσει ο χρόνος που υπάρχει για κύρωση αυτής της συμφωνίας να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την σταδιακή κατάργηση κάποιων τύπων δεξαμενοπλοίων. Ε, προφανώς επίση χρειάζεται απαραίτητη πιστοποίηση, υπάρχει μετά και η ευθύνη του κατασκευαστή. Κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει και πέρσι. Φαίνεται πως η Κομισιόν επανέρχεται σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι έχει να πει ο Επίτροπος ο κ. Φίγκελ για αυτά. Θέλω να ακούσω μάλιστα συγκεκριμένα πως η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να συστήσει ένα ταμείο για αυτή την υπόθεση. Προτείνει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκάθαρες λύσεις για μια σειρά προβλημάτων. Ελπίζω η Επιτροπή Μεταφορών και Περιβάλλοντος και χαίρομαι μάλιστα για το ότι έχουν ε, ε, βρει πλειοψηφίε σχετικέ προτάσει σε αυτέ τι επιτροπέ να πείσουν την Κομισιόν και το Συμβούλιο να εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις σχετικά για να προστατεύσουν και το περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τον Επίτροπο Φίγκελ εάν αυτή είναι η γραμμή που ακολουθείται στις διαπραγματεύσεις για τη διάσκεψη του Διεθνούς ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού και το τι θα ε, γίνει για την εφαρμογή της σχετικής σύμβασης. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το έντονο ενδιαφέρον του και συνεχές ενδιαφέρον του για τη διάλυση των πλοίων και ειδικά τον κύριο Μπλόκλαντ. Πρόκειται για μια πολύ καλή αφετηρία εδώ πέρα για περαιτέρω δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δυσφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει τον ρόλο της για την επίλυση αυτού του διεθνούς προβλήματος. Τα ζητήματα αυτά επίσης είναι επίκαιρα υπό το φως της πρόσφατης απόφασης ε, του δικαστηρίου του Μπαγκλαντές την οποία αναφέρατε. Ως αποτέλεσμα αυτής ε, της ε, απόφασης ε, όλα αυτά τα διαλυτήρια θα κλείσουν εντός δύο εβδομάδων καθώς δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Θα απαγορευτεί η εισαγωγή των επικίνδυνων πλοίων και όλα τα πλοία θα πρέπει να καθαριστούν πριν πάνε για διάλυση. Τέλος, το Μπαγκλαντές θα αρχίσει την ανάπτυξη εθνικής νομοθεσίας για τη διάλυση πλοίων που θα ευθυγραμμίζεται με τη σύμβαση της Βασιλείας. Τώρα, να έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας, στα του οίκου μας, για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Μιλάτε για τη σταδιακή κατάργηση της ε, μεθόδου της προσάραξης και της διάλυσης επιτόπου στην ακτή των πλοίων. Συμφωνώ μαζί σας. Πράγματι αυτό σημαίνει σοβαρός κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σκεφτήκαμε το ζήτημα της απαγόρευσης στην Ευρώπη της ε, προσάραξης ε, στην στρατηγική μας. Είχαμε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τέτοιας απαγόρευσης εφόσον θα ίσχυε μόνο για πλοία με σημαία κράτους μέλους και μπορούσε να παρακαμφθεί εύκολα με το να αλλάξει σημαία το πλοίο. Θεωρούμε πως θα είναι αποτελεσματικότερο να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε πως οι τεχνικές προδιαγραφές που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται όσον αφορά τις μελλοντικέ συμβάσεις του ΔΝΟ ε, να οδηγήσουν σε ασφαλή ανακύκλωση των πλοίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την κατάρτιση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και αμφιβάλλουμε ούτως ή άλλως πως ε, η μέθοδος αυτή της προσάραξης ε, θα συμμορφώνεται και με τις, γραμμέ, γραμμές που είναι αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία. Και για να σας απαντήσω, η Κομισιόν πράγματι σκοπεύει να οδηγήσει σε γρήγορη μεταφορά της σύμβασης αυτής στο κοινοτικό δίκαιο η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ήδη ξεκινήσει πολλές μελέτες και αξιολογεί τον αντίκτυπο των βασικών στοιχείων αυτή της σύμβαση. Θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει εδώ πέρα ηγετικό ρόλο και είναι υψηλή η προτεραιότητα που αποδίδουμε στο θέμα. Έτσι θα ενθαρρυνθεί η κύρωση από τρίτες χώρες και άρα θα επιταχυνθεί η θέση ενισχύ εν λόγω σύμβαση. Συμφωνώ όμω και με τις ανησυχίε που αναφέρατε στο τρίτο σας ερώτημα για το ότι δεν πρέπει να υπονομεύσουμε το κοινοτικό και εκτιμένο. Πρέπει να διατηρήσουμε τις υπάρχουσες απαιτήσει όσον αφορά το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων όταν θα μεταφέρουμε στο κοινοτικό δίκαιο τη σύμβαση του ΔΝΟ. Γι' αυτό θα συγκρίνουμε στη μελέτη μας τις διατάξεις της σχετικής σύμβασης με το κοινοτικό κεκτημένο και θέλω να τονίσω, ιδιαίτερα θα διασφαλίσουμε πως ο σχετικός, κανο... πως ο σχετικός του 2006 δεν θα υπονομευθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αγίουσο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτή η ερώτηση, όπως ε, επεξήγησε ο κύριος Μπλόκλαντ, είναι σκόπιμη αν λάβουμε ε, υπόψη το, τη διάσκεψη η οποία έχει διονοργωθεί για το Μάιο ως προς την ανακύκλωση των πλοίων. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπλόκλαντ και για το ψήφισμα που προετοίμασε. Στο ΕΛΚ θεωρούμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κακές ε, πρακτικές παροπλισμού των πλοίων. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρόταση ψηφίσματος του κυρίου Μπλόκλαντ. Στο παράρτημα 3 που είπατε και εσείς, το παράρτημα 3 μας ε, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα διότι θα πρέπει να δούμε πώς εντάσσονται αυτά τα παροπλισμένα πλοία στην Σύμβαση της Βασιλείας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι τη Σύμβαση της Βασιλείας θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη για να μην αντιφάσκουμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε επίσης και το θέμα της Διεθνούς Σύμβασης για τον ε, παροπλισμό των πλοίων. Επίσης μιλάμε για έναν μηχανισμό ε, υποχρεωτικών μέτρων ως προς τις ε, ενδοκινοτικές μεταφορές. Δεν είναι σκόπιμο να το ορίσουμε αυτό τη στιγμή που δεν έχει οριστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ποιο θα είναι το πλαίσιο ανακύκλωσης ή παροπλισμού. Τέλος, στο σημείο 15 προτρέπουμε την Επιτροπή να λάβει μέτρα σε σχέση με τη μορφή αυτή ε, αποβλήτων που αποτελεί το ίδιο το παροπλισμένο πλοίο. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη τη σύμβαση της Βασιλείας και τη σύμβαση για τον παροπλισμό των πλοίων. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τη Σύμβαση της Βασιλείας, αλλά όλη την προϋπάρχουσα νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε και τώρα δεν υπάρχει κανένας ομιλητής στο ΚΑΣΤΕΑΗ άρα ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια και από την κυρία Γιούσο και από τον κύριο Μπλόκλαντ και σε σχέση με τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα εφαρμοστεί η σύμβαση και θα συμβαδίζει με αυτή που εγκρίθηκε πρόσφατα σε σχέση με τα παροπλισμένα πλοία 10-13 του 2006. Δεν υπάρχει μηχανισμός χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή. Έχουμε ξεκινήσει με μία έρευνα για να προετοιμάσουμε τις εναλλακτικές, ή ενδυνάμει λύσεις και θα αρχίσουν οι δημόσιες διαβουλεύσεις για αυτό το θέμα. Άρα ευπρόσδεκτα θα είναι τα σχόλιά σας πάντα σε σχέση με τη σύσταση αυτού του Ταμείου Παροπλισμού των Πλοίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί. Και το επόμενο θέμα είναι η έκθεση «Λένε» για τη Λευκή βίβλο σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για την ε, παραβίαση αντιμονοπολιακής νομοθεσίας. Ο κύριος Λένε έχει το λόγο και έχουμε καθυστερήσει.